So good afternoon, colleagues. Take your seat, please. Pan Horáček také. Καλό καθίστε. We start our afternoon session. Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε τον κ. Σιμόνοβιτς, τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ διότι νομίζουμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε η Κροατία να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δυνατόν. δυνατών. Αλλά ξέρουμε ότι για να συμβεί αυτό η Κροατία θα πρέπει με αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι στο δικό χαρτοφυλάκι όπως η διαδεδομένη διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα που όπως γνωρίζουμε αυτά αποτελούν και εμπόδιο για την ανάπτυξη της χώρας σας. Ε, έχετε αρκετά δύσκολη δουλειά. Διοριστήκατε δύσκολες στιγμές για τη χώρα σας. Αλλά νομίζω ότι ήδη δείξατε αποφασιστικότητα και θάρρος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Λοιπόν, Υπουργέ, έχετε το λόγο για να προβείτε στην αρχική σας δήλωση και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις μας και οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη αυτή ευκαιρία που μου δίδετε να εκφράσω τις απόψεις της Κροατίας σχετικά με τη δικαστική μεταρρύθμιση, την μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα που λαμβάνει η χώρα και να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη της Επιτροπής για την έγκριση μιας εκθέσεως η οποία ελπίζουμε να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο τον επόμενο μήνα. Ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή διότι σε αυτές τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που κάνουμε χρειαζόμαστε ενθάρρυνση. Περνάμε μέσα από δύσκολες μεταρρυθμίσεις αρκετά δύσκολες περιστάσεις ε, λόγω της παγκόσμιας κρίσης, της ύφεση, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, παρόλο που επικρίνει κάποια πράγματα και κρίνει, κρίνει θετικά θα έλεγα γιατί μας κινητοποιεί μας οδηγεί στο να πετύχουμε τους στόχους μας, να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για το έτος, το τέλος του έτους του 2009 που είναι ο στόχος μας. Εκτιμούμε πάρα πολύ τα αρχικά προπαρασκευαστικά βήματα για την ε, επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών σαν επίσημη βάση μέσω ομάδας του σχεδίου της Συμφωνίας Προσχώρησης. Όσον αφορά το δικαστικό σύστημα στην Κροατία, μπορώ να ανακοινώσω ότι πάντα ε, θεωρούμεθα θεωρούσαμε ότι αυτό ε, ήταν εμπόδιο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αλλά δηλώνω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τον μονόλογο, θα πω μερικά λόγια μόνο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς. Διορίστηκα υπουργό Δικαιοσύνης πρωτετραμίνου στις 6 Οκτωβρίου πέρσι. Έγινε μια φρικτή δολοφονία στην πόλη του Ζάγκρεμπ, στην ποτέουσα της Κροατίας. Μια νέα γυναίκα, 26 ετών, δολοφονήθηκε στο κέντρο της πόλης, 100 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα και υπήρχαν σοβαρές υπόνοιες ότι ήταν θύμα του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο οργανωμένο έγκλημα έκανε επίδειξη δύναμης και ατιμορρησίας. Αυτή η δολοφονία οδήγησε στην αλλαγή του Υπουργού Εσωτερικών, Υπουργού Δικαιοσύνης και του Διευθυντή της Αστυνομίας. Και ανέλαβα ένα καθήκον να διοργανώσω μια αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και να επιταχύνω τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ε, λύθηκε το ζήτημα επιτυχώς, αλλά ανακαλύψαμε ότι η κυρία αυτή δεν ήταν θύμα του οργανωμένου εγκλήματος, εξηχνιάστηκε, αλλά ενός ψυχοπαθούς αστέγου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάποιος βαθμός οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι τόσο ομό και άγριο όπως είχαμε φανταστεί το οργανωμένο έγκλημα αλλά παρόλα αυτά έχουμε αποτελεσματικότατο σύστημα που θα καταπολεμά τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα στο οποίο εντάσσονται ειδικέ αστυνομικέ δυνάμει, ειδικό τμήμα του Γενικού Εισαγγελέα και σε 10 μέρες περίπου θα έχουμε και ειδικά δικαστήρια, ειδικά τμήματα δικαστηρίων που θα είναι υπεύθυνα για την καταδίωξη και εκδίκαση εγκλημάτων διαφθοράς και περιπτώσεων πράξεων του οργανωμένου εγκλήματος. Εισαγάγαμε επίσης μια και πολλές καινοτομίες μάλλον στο σύστημά μας που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Εισαγάγαμε ένα άρθρο το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα για κάθε άτομο που καταδικάζεται για διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα να υποτίθεται, να θεωρείται ότι όλη η περιουσία του αποκτήθηκε παράνομα και κατάσχεται η περιουσία αυτού του ατόμου. Αυτό το άρθρο μας δίνει δυνατότητα να κατάσχουμε στοιχεία ενεργητικού που διαβάστηκαν σε τρίτα πρόσωπα, σε συγγενείς ή τρίτα πρόσωπα, αν ο εισαγγελέα η αρχή μπορεί να αποδείξει ότι αυτό έγινε για να αποφευχθεί ε, κατάσχεση παρανόμως αποκτηθήσας περιουσίας. Να αναφερθώ ακροθυγώς σε θέματα που απτονται της δικαστικής μεταρρυθμίσεως. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν θέλουμε απλώς γραφειοκρατικά να πετυχαίνουμε στόχους και να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, να πετύχουμε πρόοδο στην μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου και πάνω σε αυτό έχω να τονίσω τρία βασικά καθήκοντα που θέλουμε να εκτελέσουμε. Θέλουμε δικαιοσύνη που θα είναι ταχεία, αμερόληπτη και προσβάσιμη τη πάση. Όσον αφορά την ταχύτητα, αλλάξαμε αρκετούς νόμους, διαδικαστικό δίκαιο, για το αστικό δίκαιο, για το ποινικό δίκαιο, ε, για τα διοικητικές, διοικητικές κυρώσεις για να επιταχυνθούν οι διάφορες διαδικασίες. Έχουμε εξορθολογήσει το δίκτυο των δικαστηριών μας και μειώσαμε στο μισό το δίκτυο αυτό, ούτω ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους λίγους πόρους που διαθέτουμε, τους δικαστές μας, παραγωγικότερα. Τώρα, επίσης, υπήρξαμε επιτυχείς όσον αφορά το να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο, να καλύψουμε υποθέσεις που είχαν καθυστερήσει, είχαν μείνει πίσω. Κάθε χρόνο μειώνεται ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν ε, καθυστερήσει. Έχουμε τρίγωνο μεταξύ Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Προέδρων των διαφόρων δικαστηρίων και του Υπουργού του υποφωνωμένου και στο τρίγωνο αυτό έχουμε, συμφωνήσει ένα πρόγραμμα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και ο πρόεδρος κάθε δικαστηρίου ελέγχεται κατά πόσο υπήρξε επιτυχή στη διαχείριση του δικαστηρίου του. Αν τελικά καλύπτει τη χρονική υστέρηση όσον αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων, όσον αφορά την αμεροληψία, εισάγουμε ένα σύστημα ε, επιλογής και προαγωγής δικαστών βάσει της αξίας τους και ξεκινά κρατική σχολή δικαστών Μέσω διαγωνισμών θα γίνει τη εισαγωγή, μέσω γραπτών εξετάσεων και μετά την αποφύτιση. Για την αποφύτιση μάλλον χρειάζονται πάλι γραπτές εξετάσεις βάσει βαθμολογίας. Λοιπόν, βάσει της βαθμολογίας καταρτίζεται κατάλογος, εθνικός κατάλογος υποψηφίων για τα δικαστήρια. Έχουμε επίσης κατάλογο κενών θέσεων κάθε χρόνο στα δικαστήρια και για το ε, γραφείο του Ισαγγελέως και αυτοί που έχουν την καλύτερη βαθμολογία είναι εκείνοι που μπορούν να διαλέξουν που θα εργαστούν στην Κροατία ως δικαστές ή ως εισαγγελείς. Να πω κάτι όσον αφορά την προσβασιμότητα της πάση. Από φέτος το Φεβρουάριο έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα ελεύθερης νομικής αρρωγής και έτσι ο καθένας, ανεξάρτητα της κοινωνικής και οικονομικής του θέσης, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δικαστήρια και θα μπορεί επιτυχώς να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, professor. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Οι συνάδελφοι ο κύριος Σβόμποντα που είναι και ο εισηγητής για την Κροατία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζω τον κύριο Υπουργό. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και πριν από δύο εβδομάδες στο Ζάγκρεμπ και ο επαγγελματισμός και αποφασιστικότητά του να κάνει αυτά που λέει με έπεισαν. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό κάτι που δεν συνέβαινε με άλλες περιπτώσεις αυτών που σας ε, διόρισαν. Εγώ χαίρομαι που σας διορίσαν, αλλά αυτό δεν ισχύει για άλλες περιπτώσεις. Με μια σειρά θεμάτων θέλω να ασχοληθώ. Η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στον δικαστικό τομέα. Προφανώς δεν είναι εύκολος ε, τομέας. Υπάρχουν αντιστάσεις. Επισκεφθήκαμε με τον κύριο Μπροντζάτο τα δικαστήρια στην Κροατία διαπιστώσαμε ότι ναι μεν υπήρχε βούληση να ε, γίνουν αλλαγέ, απ' την άλλη φοβόντουσαν να προχωρήσουν γρήγορα. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα πολλοί επενδυτές που έρχονται και μας λένε ότι έχουν προβλήματα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, από τα διοικητικά μέτρα, από τον προστατευτισμό των ντόπιων εις βάρος των ε, ξένων επενδυτών. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήταν σημαντικό να δείτε το θέμα αυτό, γιατί είναι κακό για την Κροατία. Προφανώ είναι κακό και για του ε, ιδιώτες επενδυτέ, αλλά είναι κακό να μην υπάρχει ανταγωνισμό για την Κροατία και να μην έρχονται επενδυτέ. Και στην... δεν είναι μοναδική κατάσταση στην Κροατία, το ξέρουμε και στι δικέ μα χώρε. Ακούγεται, υπάρχει το... η αίσθηση ότι υπάρχει όλο το σύστημα ακόμα αντιμετωπίζει δυσμενώς τους ξένους. Το γεγονό, για παράδειγμα, ότι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο μια επιχείρηση πρέπει κάποιο να μιλάει κροατικά, που είναι καλό, ερμηνεύθηκε όσο ότι κάποιο πρέπει να, είναι, να έχει την κροατική υπηκότητα. Επίση, μπορείτε να μα πείτε και δύο λόγια για την ε, συνεργασία σα με το Διεθνέ Ποινικό δικαστήριο για τη Ιουγκοσλαβία. Υπάρχουν ακόμα καταγγελίες και παράπονα για την ε, παράδοση κάποιων εγγράφων. Θα ήταν σκόπιμο να ξεκαθαριστούν τα πράγματα αυτά. Μήπως μπορείς να ενημερώσει την Επιτροπή για το πώς έχουν τα πράγματα. Κάποια κακά νέα στις εφημερίδες έλεγαν, κοιτάξτε να δείτε, δεν συνεργάζεται πλήρως η Κροατία, άρα θα πρέπει να επανεξετάσουμε το χρονικό ορίζοντα που είπε ότι μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ελπίζω τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν γρήγορα, αλλά θα μπορούσατε να μας πείτε πέντε πράγματα κι εσείς για το πώς βλέπετε την κατάσταση. Αυτά. Τελειώνω πρόεδρε για να δώσω και στους συναδέλφους την ευκαιρία να μιλήσουν. Thank you, Η Doris Σπακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ χαίρομαι που ε, σας ξαναβλέπουμε με διαφορετική ιδιότητα. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια ε, είχατε βέβαια πολλά αξιώματα στην Κροατία. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι και εγώ πως και ο Χάνες που σας βλέπω με τη σημερινή σας ιδιότητα. Αυτά που μας είπατε μας καθιστούν ιδιαίτερα αισιόδοξου για το ότι η δικαστική εξουσία στην ε, Κροατία θα εξελιχθεί κάτι που είναι απαραίτητο για να καταστεί η Κροατία μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι και προς όφελος της ε, Κροατίας. Ε, αυτό που κάνουμε με την Κροατία το Συμβούλιο δεν το έπραξε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και γνωρίζουμε πλέον ότι δεν είναι δυνατόν ούτε για τη χώρα αλλά ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχόμεθα χώρες οι οποίες δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στον τομέα αυτό. Το να κάνει κανείς τα πάντα αυτό είναι δύσκολο. Είναι όμως σημαντικό να γίνουν σημαντικά άλματα. Θεωρώ λοιπόν ότι εσείς ελέγχετε την κατάσταση και πιστεύω ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον δικαστικό τομέα. Υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις ε, που δεν ε, έχουν εξεταστεί, σορεύονται εδώ και χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για τους ενδιαφερόμενους και πολλοί εξ αυτών έρχονται σε μένα για να τους βοηθήσω. Αλλά και εγώ τι να κάνω. Αυτά είναι θέματα των οποίων πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι σημαντικό να υπάρξει κάποια βελτίωση. Το βασικότερο όμως είναι αυτό που είπε στο τέλος ο Γιωχάνης. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι εντωμεταξύ προβάλλεται το επιχείρημα της ε, μη πλήρους συνεργασίας με το ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Το θέμα δεν είναι ε, ότι δεν έχουν εκδοθεί οι καταζητούμενοι. Αυτό συνέβη, υποδειγματικά μάλιστα, και γι' αυτό εμείς είμαστε υπερήφανοι. Το πρόβλημα είναι ότι από ό,τι φαίνεται, για να παραδοθούν οι κατηγορούμενοι, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αποδείξεις οι οποίες βρίσκονται κάπου στα αρχεία της Κροατίας. Τουλάχιστον αυτό ισχύει το κ. Μπράματς και η δική σας η κυβέρνηση λέει, ισχυρίζεται ότι ε, καταβάλει προσπάθειες και ψάχνει στοιχεία αλλά δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μπράμας και εκείνος ε, δεν ε, είδε συγκεκριμένα πράγματα αλλά ε, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν μάρτυρες που είδαν αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης το 2005. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά αλλά γνωρίζουμε όλοι μας ε, ότι το θέμα αυτό επιβαρύνει τις διαπραγματεύσεις. Αν λοιπόν μπορείτε να κάνετε κάτι έτσι ώστε να αμβληνθούν κατά τη οι κατηγορίες ή αν θέλετε τα γεγονότα ε, εφόσον δεν υπάρχουν ε, αποδείξεις να χαρακτηριστούν ως παροχημένα. Αν όμως υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που κάπου έχουν σωρευθεί, τότε πιστεύω ότι η κυβέρνηση της Κροατίας πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δοθούν αυτές οι αποδείξεις. Νομίζω τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Η έκδοση ήταν το χειρότερο που μπορούσε να γίνει και γι' αυτό θεωρώ ότι αν κύριε Υπουργέ ε, μπορείτε να παρουσιάσετε κάποια στοιχεία ε, τα οποία θα κρυθούν ως αποδείξεις, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό. Έχετε προβλήματα με τους ε, γειτονές σας, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχετε και προβλήματα με το ποινικό δικαστήριο. Εγώ ήθελα να πιστεύω ότι το θέμα έχει λήξει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει λήξει και γι' αυτό το λόγο θέλω να ελπίζω ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια. Κύριε Σεντριβάνη από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, κύριε Σιμωβίτς, πρέπει να σας ε, συγχαρώ για, την, ε, για το βιορισμό σας. Πολλά καλά νέα έχουμε από τη δικαιοσύνη στην Το καλύτερο είναι η τοποθέτησή σας εσύ εκεί. Κάτι το είπε, το, το δήλωσε και η Βέσνα Πόσιτς, η ηγέτη της αντιπολίτευσης που χαιρέτησε την επιλογή σας στη θέση αυτή. Καλό νέο λοιπόν. Βεβαίως, Ακούσαμε καλά λόγια για τις ε, προθέσεις σας. Θέλουμε ωστόσο και πράξεις τώρα. Πράξεις που θα υλοποιηθούν σύντομα και συγκεκριμένα βήματα. Είσαστε ένα σύμβολο, μία υπόσχεση, αλλά η υπόσχεση πρέπει να τηρηθεί. Δεύτερο θέμα, το είπαν οι συνάδελφοι. Ο κ. Πλάμετς πρόσφατα δήλωσε ότι η Κροατία δεν συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Δικαστήριο για τα Εγκλήματα στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Πόσο γνωρίζω, το μόνο πρόβλημα είναι το μητρό του πυροβολικού που δεν υπάρχει ακόμα. Στοιχεία, τα στοιχεία αυτού του μητρώου πού είναι, χάθηκαν όντως, τι προτίθεστε να κάνετε για να τα βρείτε. Πώς έχει η κατάσταση. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στην ε, ε, εκκρεμή. Επίσης, τι γίνεται με την ε, μεθοριακή διένεξη με την ε, Σλοβενία. Πολλοί από εμάς εξεπλάγημεν από την, ε, το εμπάργο στη Σλοβενία. Εμείς πιστεύουμε εγώ προσωπικά είμαι τελείως αντίθετος με οποιαδήποτε προσπαθία να χρησιμοποιηθείτε ως όμοιροι για, η διεύρυνση μάλλον χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επίλυση των μεθοδιακών αυτών ε, θεμάτων. Γιατί η διεύρυνση είναι ένα μείζον εγχείρημα της ε, ε Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπόκειται σε ε, εθνικές απαιτήσει. Βεβαίω πρέπει να υπάρξει ευελιξία και από τι δύο πλευρέ. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση τη κυρία Σιμόνοβιτ για να δείξει ευελιξία από πλευρά σα. Το ίδιο περιμένουμε και από την σλοβενική πλευρά. Και μια επικοδομητική συμπεριφορά από πλευρά σα. Thank you. And finally in this first round of questions, Mr. Horacek. Ja, danke schön. <clears throat> Ähm, es wurde nach den, nach den äh, äh, Ο Ιβάνα Χόντα και ο Ιπο Πουκάνιτς είπαν ότι όχι μόνο η δικαστική μεταρρύθμιση αλλά και η αστυνομική μεταρρύθμιση επίκυνται και ότι θα ε, συσταθούν επιπρόσθετα δικαστήρια. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας πείτε λίγα λόγια επ' αυτού, διότι άλλο πράγμα η δικαστική μεταρρύθμιση και άλλο η αστυνομική. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι γίνεται στην Τσεχία και εκεί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Κατόπιν έχω άλλο ένα ερώτημα που αφορά στο νέο νόμο για τα γήπεδα του γκολ. παρατηρούμε, ξέρετε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται τεράστιες εκτάσεις ε, για γήπεδα γκολφ, ε, κυρίως ε, στις παραλίες, αλλά και στην ενδοχώρα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχω επισκεφθεί επανειλημμένα την Κροατία. Ξέρω ότι η Κροατία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον τουρισμό. Το θέμα όμως είναι μήπως με τη δημιουργία αυτών των γηπέδων του γκολφ θίγονται τα συμφέροντα των Κροατών. Ίσως ε, οι εκτάσεις αυτές ε, που θα χρησιμοποιηθούν για γήπεδα ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για οικολογικές καλλιέργειες, βιολογικές καλλιέργειες, για την παραγωγή κρατού, κρασιού, για μπέλια. Ίσως θα μπορούσατε να πείτε και από αυτού δύο λόγια. Δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Υπουργός παίζει γκολφ. Ε, φαντάζομαι θα το ξέρει όμως το θέμα και θα μπορεί να τοποθετηθεί από αυτού. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω εν συντομία να αναφερθώ σε όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν. Ε, να απαντήσω στον κύριο Σβόμποντα σχετικά με τις επενδύσεις και τον προστατευτισμό. Η Κροατία ενδιαφέρεται και πολύ μάλιστα για ξένες επενδύσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι χωρίς αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των ενδιαφερομένων, είτε είναι Κροάτες, είτε είναι αλλοδαποί, είναι σημαντικό. Πρέπει να στατεύονται όλοι οι επενδυτές. Έτσι θα προσελκύσουμε κεφάλαια. Τώρα, οι προσπάθειες για την επίτευξη αμεροληψίας στα δικαστήριά μας. Να σας δείξω ότι κάναμε ένα μέτρο. Περίπου σε μία εβδομάδα θα βάλουμε σε ιστοσελίδα όλες τις αποφάσεις το ανωτά του εμπορικού μας δικαστηρίου. Τίποτα δεν θα διαγράφεται. Θα αναφέρονται πλήρως οι αποφάσεις. Όνομα δικαστού, όνομα επιχειρήσεως, είτε είναι κρατική επιχείρηση είτε ξένη. Και θα μπορεί κανείς να ερευνά τις βάσεις δεδομένων μέσω υπολογιστού και έτσι όλοι θα μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει η αδίποτε απόπειρα να υποστηριχθεί συγκεκριμένο, μεροληψία δηλαδή, αν έχω αντιμετωπιστεί ισότιμα οι ξένοι ή όχι. Θα είναι εύκολα προσβάσιμες οι πληροφορίες. Έτσι θα διαπιστώνεται η αμεροληψία μας και τα, κατά πόσο τα εμπορικά δικαστήρια είναι αμερόληπτα ή όχι. Και θέλουμε να είναι όχι μόνο ανεξάρτητα δικαστήρια αλλά και αμερόληπτα. Πολλοί ερώτησαν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία και θα ήθελα να αναφερθώ σε θέματα συνεργασίας με την εισαγγελία όσον αφορά αυτά τα ημερολόγια του πυροβολικού και τα διάφορα έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του κ. Μπράμιτς. Μας ανησυχεί όλους ιδιαίτερα στο θέμα. Μίλησα με τον κύριο Σαγγελέα, τον κύριο Μπράμιτς, χτες το βράδυ και συνεχίζεται η συζήτησή μας την Παρασκευή. Πράγματι, θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οι εκκρεμότητες πώς θα επιληθούν. Αυτό είναι κάτι που δυσαρεστεί τον κύριο Μπράμιτς. Δύο πράγματα μάλλον. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποια έγγραφα που λείπουν και του χρειάζονται για τη δικογραφία. Δεύτερον, δεν παίρνει απάντηση από την κυβέρνηση της Κροατίας κατά πόσο αυτά τα έγγραφα έχουν παραχθεί και λείπουν ή κάποια έγγραφα δεν υπήρξαν ποτέ διότι κάποιες μονάδες δεν συμμορφωνόταν πλήρως με τους κανόνες. Για τον κύριο Μπράμερτς. Με τον κύριο Μπράμερτς τελειώνουμε την ανάλυση. Για κάθε έγγραφο που τον ενδιαφέρει γίνεται εξέταση. Καταρτίστηκε κατάλογος εγγράφων από μια συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων που έλαβε χώρα στο Ζάγκρεπ. Κάλεσα προσωπικά τον κύριο Μπράμερτς να έρθει στο Ζάγκρεπ να καθαριστούν αυτά τα θέματα εντόπισε 33 έγγραφα τα οποία υποτίθεται ότι υπήρχαν και εμπεριείχαν σημαντικά στοιχεία για τον εισαγγελέα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι έλεγχος κατά πόσο αυτά τα 33 έγγραφα υπήρχαν ή δεν υπήρχαν Θα ξεκαθαριστεί λοιπόν το θέμα της 15 Φεβρουαρίου. Για τα έγγραφα που υπήρξαν και δεν είναι τώρα προσβάσιμα, θα κανονίσουμε ποιος θα είναι υπεύθυνο, ποιο πρέπει να τα έχει την προστασία του. Αν έχει ετοιμαστεί ένα έγγραφο, κάποιος κάποτε θα έχει στην κατοχή του αυτό το έγγραφο. Για καθέναν που ήταν ο τελευταίος που νομίμως ήταν κάτοχος του εγγράφου, προβλέπεται υποχρέωση είτε να παρουσιάσει και να υποβάλει ένα έγγραφο στην κρατική κυβέρνηση και η κρατική κυβέρνηση με τη σειρά της να το υποβάλει στο δικαστήριο, είτε αυτός ο άνθρωπος που ήταν ο τελευταίος κάτοχος του εγγράφου θα υποστεί τις νομικές συνέπειες. Για να ξεκαθαριστεί η θέση της Κροατίας και της εισαγγελία. ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε ένα κοινό έγγραφο που θα είναι έγγραφο της κυβέρνησης Κροατίας και της Ισαγγελίας. Και το έγγραφο αυτό θα αναφέρει επακριβώς ότι η Κροατία έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αστυνομικά έγγραφα, επίσης για την ίδια στρατιωτική επιχείρηση και υπάρχουν και άλλα συναφή έγγραφα που αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά υπάρχουν κάποια έγγραφα που ακόμα λείπουν. Θα απαριθμούνται λοιπόν τα έγγραφα που λείπουν. Και θα τονίζετε ότι αυτά τα έγγραφα υπήρχαν αλλά τώρα λείπουν και θα δίνονται διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα ώστε να ξεκαθαριστεί ποιος ήταν ο κάτοχος αυτού του εγγράφου, με ποια διδοχή σειρά και να υποστούν τις νομικές συνέπειες τα άτομα εκείνα που ήταν οι τελευταίοι κάτοικοι, ε, κάτοχοι των εγγράφων που ζητάει ο κ. Μπράμετς. Τώρα το ερώτημα της κυρίας Πακ. Δεν μας πειράζει να συμμορφωθούμε τις απαιτήσει του κεφαλαίου 23. Είναι καλό για την Κροατία. Είναι χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για μεταρρυθμίσεις που ούτως ή άλλως χρειάζονται. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα ήταν κάτι που χρειαζόταν η Κροατία και θα το κάνουμε. Και το κεφάλαιο 23 δεν μπορεί παρά να μας βοηθήσει σχετικά με αυτό το σκοπό. Καμιά φορά ως υπουργό Δικαιοσύνης είναι για μένα πιο εύκολο να πω ότι δεν είναι μονολογικό, αλλά επίσης είναι και απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καμιά φορά δεν καταχρώμαι, αλλά κάπως χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα του κεφαλαίου 23. Όσον αφορά άλλα ζητήματα που έθεσε ο κ. Σαντιβάνη Συμφωνώ απολύτω. Χρειαζόμαστε πράξεις. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Φτάνουν οι υποσχέσεις. Τι να πω εγώ για τις συγκεκριμένες πράξεις μου. Επιφέραμε οργανωτικές βελτιώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Για πρώτη φορά, δεν το είχαμε αυτό, για πρώτη φορά θα έχουμε ειδικέ αστυνομικέ μονάδε επιφορτισμένε με την καταπολέμηση τη διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος Υπάρχουν τώρα και άλλο ερώτημα ετέθη για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Αυτές οι μονάδες αποκτούν ε, προχωρημένη τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία ε, ο εξοπλισμός τους ήδη λειτουργεί, ήδη μπορεί να κινηθούν αυτές οι μονάδες. Όσον αφορά το ειδικό τμήμα της εισαγγελία υπήρχε, αλλά ενισχύθηκε. Για πρώτη φορά, σε περίπου 10 μέρες, ε, θα έχουμε 60 δικαστές που θα είναι ειδικοί δικαστές για τα τμήματα των δικαστηρίων, που θα είναι φορτισμένοι κυρίως για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις υποθέσεις. Και έχουμε θεσπίσει ένα κανόνα ότι υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να εξετάζονται πρώτα, μετά από 7 ημέρες, αφού έχει υποβληθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Και για αυτές τις υποθέσεις κάθε μήνα ένας δικαστής που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση θα πρέπει να υποβάλει στον πρόεδρο του δικαστηρίου σχετική έκθεση. Ε, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος ούτε ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου είναι ικανοποιημένος με κάποιους πρόεδρους δικαστηρίων διότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί ή διότι έχουν δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Έχω απολύσει τρεις προέδρους δικαστηρίων το τελευταίο τετράμινο. Το ίδιο ισχύει για τεσσάρους διευθυντές φυλακών στην Κροατία λόγω διαφόρων προβλημάτων και ελλείψεων στο έργο που επιτελούσαν. Αυτά είναι τα πλέον πρακτικά μέτρα τα οποία μπορώ να παριθμίσω για να σας δείξω ότι πράγματι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά και προσβλέπω σε περαιτέρω στοιχεία να δούμε κατά πόσο τελικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί επηρεάζουν τη χρονική καθυστέρηση που είχαμε διαπιστώσει υποθέσει. Εγώ πιστεύω θα αρχίσουμε να καλύψουμε τη χρονική στέρηση. Και η αλλαγή τη νομοθεσία και η μεγαλύτερη πίεση επί των πρόεδρων των δικαστηρίων θα δώσουν αποτελέσματα. Διότι πρέπει να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα δικαστήρια. Όχι να είναι απλώ καλοί δικαστέ, να είναι καλοί manager. Τόσο αφορά τη Σλοβενία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό το θέμα βλάπτει και τη Σλοβενία και την Κροατία. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να βρει λύση. Εκ μέρους της Κροατίας μπορώ να πω ότι θα παράσχουμε όλα τα αναγκαία εχέγγυα στη Σλοβενία ούτω ώστε να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες της. Το μόνο όριο είναι ότι η Κροατία δεν μπορεί να απεμπολίσει την επικράτειά της, τα δικαιώματά της αυτά και απαιτεί την εφαρμογή νομικών κανόνων όσον αφορά τον καθορισμό των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Όσον αφορά οποιασδήποτε άλλες ανησυχίες της Σλοβενίας, εμείς θα προσπαθήσουμε να τις λάβουμε υπόψη και να θεωρήσουμε ότι δεν είναι απλώς γειτονική μας χώρα, αλλά είναι γειτονική χώρα με την οποία είχαμε ιστορικά έξοχες σχέσεις και είναι κρίμα τώρα να έχουμε αλλαγές απόψεων στην κοινή γνώμη και επιδείνωση των σχέσεων. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από πλευράς Σλοβενίας και Κροατίας αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες Όσον αφορά τώρα το τελευταίο ζήτημα σχετικά με τα γήπεδα του γκολφ ψηφίστηκε ο νόμος για τα γήπεδα του γκολφ στην Κροατία δεν έχουμε ούτε ένα γήπεδο του γκολφ ακόμα ποια ήταν η ιδέα για τέσπιση του νόμου να δώσουμε κίνητρα ούτω ώστε να δημιουργηθούν γήπεδα του γκολφ ακούστηκαν όμως και κάποια σχόλια ότι ο τρόπος η κυβερνήση πήγαινε τα πράγματα πολύ μακριά, αλλά διεξάγεται στο εσωτερικό της χώρας σχετικός διάλογος εσωτερικός κυβερνήσεως. Thank you. Ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος, ο κ. Πριμπέτιτς. Κύριε Υπουργέ, Σύντομα, θα σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε για τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη μάχη κατά της διαφθοράς, την μεταρρύθμιση της δικονομίας. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω κάποια σημεία που ε, ε, θα μπορούσε να μειώσει τις, ε, ε τις παρανοήσεις η Κροατία, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, έχει φυσικό προορισμό την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα για να ολοκληρωθεί ο ευρωπαϊκός χώρος και να συμμετάσχει η χώρα στη δυναμική και την ανάπτυξή μας. Ωστόσο θα πρέπει κάποιες παρανοήσεις, να τις, κάποιες παρεξηγήσεις να τις διαλευκάνουμε. Και συνάδελφοι και εγώ υπογραμμίζουμε την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με το ποινικό δικαστήριο για τα εγκλήματα της πρώην, στην πρώην Ιουγκοσλαβία με διάφανο τρόπο και να επιτρέψουμε με τη διαφάνεια να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις που ανέφερα. Δεύτερον, να αντιμετωπίσετε και την ιστορία. Ε, ο Αριστίδ Μπριάν, ένας Γάλλος πρόεδρος από τους σημαντικότερους, είχε πει ότι η περιοχή αυτή είχε μια πολύ αναταραγμένη ιστορία πολλές μειονότητες, ε, υπήρχε η Ιταλική μειονότητα η οποία υπέστη τις συνέπειες του πολέμου και δίωξη κατά βάση με κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Θα περίμενα να υπάρξει μια προσεκτική αντιμετώπιση της περιουσίας των μειονοτήτων αυτών, ούτως ώστε να ξεπεραστεί ε, αυτό το ζήτημα το ζητάμε και για άλλες χώρες, π.χ. την Τουρκία σήμερα το πρωί. Επιπλέον με τους φίλους από τη Σλοβενία θα πρέπει να βρείτε και ένα σημείο συνεννόησης. Τώρα, το ότι δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ για το που φτάνουν τα χωρικά ίδρυτα του Πυράν ε, ε, για τον μέσο Ευρωπαίο είναι ακατανόητο. Τώρα δίπλα είναι το πυράν και το πυράκι. Τώρα, άμα πάνε 5 μέτρα εδώ, 5 μέτρα εκεί, δεν νομίζω ότι αυτό είναι μείζον ζήτημα. Ο περισσότερο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν το καταλαβαίνουν. Και το λέω σε εσά, το λέω και στου Σλοβαίνου φίλου. Βρείτε ένα σημείο συνεννόηση, σα φύγει το ζήτημα αυτό από πρόσκομα στην ενταξιακή διαδικασία. Γιατί όταν ακούσαμε ότι ε, δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό λόγω τη ε, παρεμπόδιση πρόσβαση στη θάλασσα, Πραγματικά οι περισσότεροι δεν καταλάβαμε το πρόβλημα. Προσπαθήστε λοιπόν να το δείτε και ας προσπαθήσουμε να κλείσουμε τα υπόλοιπα 13 κεφάλαια για να μπορέσετε να έρθετε στην Ένωση όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας Ευρωπαίων, νομίζω, να έρθει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις. Απαντήσετε εν μέρη στη μία. Είπατε για την ανάγκη βελτίωση του δικαστικού σώματος. Ένα κομμάτι του είναι η ικανότητα των δικαστών να καλύψουν και να δώσουν, να κρίνουν όλες τις αποφάσεις, όλες τις υποθέσεις που έχουν μπροστά τους. Αποτέλεσμα, μεγάλες καθυστερήσεις Είπατε ότι για κάποια εγκλήματα διαφθοράς θα επιταχύνετε την διαδικασία. Αλλά για τους υπόλοιπους πολίτες τι γίνεται. Έχετε τη δυνατότητα να διορίσετε καλούς δικαστές για να προχωρήσει το σύστημα. Δεύτερον, τι κάνετε με προγράμματα προστασίας μαρτύρων. Έχετε οργανωμένο έγκλημα στη χώρα σας. Όταν έχει κανείς να αντιμετωπίσει οργανωμένο έγκλημα, το βασικό πρόβλημα είναι πώς θα πάρεις κάποιον μάρτυρα πείθοντάς τον να ε, ε, μαρτυρήσει προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα. Μια ερώτηση κι εγώ. Οι μεθοριακές διαφορές. Είπατε ότι θέλετε τη βοήθεια τη Ένωση. Εγώ ρωτώ πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήρθε ο επίτροπος Ρεν στην Κροατία πήγε στη Σλοβενία πριν από δύο εβδομάδε. Υπήρχε μια πρόταση να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του Αχτισάρη. και είναι η άποψή σα για την αντιμετώπιση του προβλήματο όπω περιέγραψε. Ευχαριστώ. Now Να απαντήσω. Για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων των ατόμων η περιουσία των οποίων είχε κατασχεθεί, είχε δημευθεί μάλλον ε, ε, σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Το εξετάζουμε. Μάλιστα, το συνταγματικό δικαστήριο αμφισβήτησε ένα, μια νομική διάταξη για να διασφαλιστεί ότι η περιουσία του καθενός ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση, Κροάτη ή άλλου, ε, εμπλέκεται. Υπάρχει και η απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου Τώρα περιμένουμε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Μετά από την απόφαση αυτή θα εξετάσουμε κατά πόσο χρειάζεται να υπάρξει νέος νόμος για να τηρηθεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την επιστροφή περιφερειών. Περιμένουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που αναφέρθηκε ως το δικαίωμα της Σλοβενίας να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Θέλω να σας διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχουν νομικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση της Σλοβενίας στη θάλασσα. Στηρίζεται στην διεθνή νομοθεσία και η απόφασή μας είναι να επιτρέψουμε πλήρη πρόσβαση της Σλοβενίας στην, ε, ε, στην ανοιχτή θάλασσα και δεν αφορά μόνο σκάφη με σημαία Σλοβενίας αλλά σκάφη με οποιασδήποτε σημαία που θέλει να φτάσει στο λιμάνι, σε λιμάνι της Σλοβενίας. Επίσης επιτρέπει την, την πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα ε, πολεμικών σκαφών και, αεροπλανοφόρα να είχε η Σλοβενία δεν θα μας πείραζε να επιτρέπουμε την πρόσβαση της ε, Σλοβενίας στην ανοιχτή θάλασσα από τα χωρικά μας ύδατα. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι κάτι άλλο. Η Σλοβενία θέλει να έχει άμεση πρόσβαση με, την, το ανοιχτό πέλαγος, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ανάμεσα υπάρχει, ανάμεσα στα χωρικά ύδατα της Σλοβενίας και την ανοιχτή θάλασσα υπάρχουν τα χωρικά ύδατα της Κροατίας. Δεν είναι ότι δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Έχει λιμάνι και μεγάλο κιόλα. Δεν υπάρχει πρόσβαση λοιπόν της Σλοβενίας στην ανοιχτή θάλασσα. Αν ανησυχεί γι' αυτό η Σλοβενία, η κυβέρνησή μας είναι έτοιμη να δώσει ό,τι εγγύηση χρειάζεται για την πρόσβαση της Σλοβενίας στην ανοιχτή θάλασσα στα διεθνή ύδατα δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βοήθεια από την Επιτροπή, την Διεθνή Ένωση, από τον Αχτισάρη, τον Μπαντεντέρ, κάποιον τέλο πάντων. Εμείς καλωσορίζουμε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση και υποστήριξη για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες μεταξύ των δύο χωρών. Η μέθοδος ωστόσο απόφασης της γραμμής των συνόρων δεν είναι πολιτικό θέμα, αλλά νομικό. Ιστορικά, δύο τρόποι υπάρχουν επίλυσης των διαφορών. Το ένα είναι ο συμβιβασμός και το άλλο είναι η επικυριαρχία. Ο συμβιβασμός σημαίνει πολιτικές διαπραγματεύσεις, επικυριαρχία σημαίνει ο δυνατότερος ή αυτός που έχει περισσότερους συμμάχους επιβάλλει τη βούλησή του στον άλλο. απετέλεσε ιστορικό γεγονός της διεθνής σχέσης και, την διεθνή, ε, και το διεθνές δίκαιο το γεγονός ότι όταν τα κράτη δεν συμφωνούν για ένα θέμα να επιλύουν το θέμα αυτό διανομικά μέσω δικαστηρίων. Είτε το δικαστήριο αυτό στηρίζεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για, την, για το δίκαιο του, των θαλασσών, το, το δικαστήριο του Αμβούργου ή ε, το Διεθνές Δικαστήριο είναι αδιάφορο. Πρόκειται ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, για, δύο περιπτώσεις για όργανα που βασίζουν την επίλυση αμφισβητούμενων διαφορών. Και θέλουμε αυτά τα όργανα να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις κατά τις οποίες πολιτικά δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτικής λύσης. Όποια προσπάθεια βοήθειας ε, ή υποστήριξη από διαμεσολαβητή που θα βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε ότι θα έχει το δικαίωμα η Σλοβενία για πρόσβαση στα διεθνή ύδατα και θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε ταυτόχρονα την μεθοριακή γραμμή ε, την μεθοδιακή γραμμή πολιτικά θα ήταν θετικό και για τις δύο χώρες νομίζω. Η ικανότητα τώρα αντιμετώπισης των δικών από τα δικαστήρια. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε την ικανότητα των δικαστηρίων να αντιμετωπίσουν την δίκη και να εξασφαλίσουμε ότι θα μειωθούν οι καθυστερήσεις. Έχουμε ετήσια πρόοδο για την μείωση των διαδικασιών Οι καθυστερήσεις είναι όλο και πιο σύντομες και εμείς προχωρούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από πολλές οπτικές γωνίες. Πρώτον, εισάγουμε, υιοθετούμε νομοθεσία που επιταχύνει τη διαδικασία, την ποινική διαδικασία, τις δικαστικέ διαδικασίες. Αλλάξαμε όλα, όπως σας είπα, αλλάξαμε όλα τα δικονομικά μας δίκαια και την αστική και την ποινική και τη διοικητική δικονομία και αυτέ οι αλλαγές ε, δείχνουν τα αποτελέσματα. Οι δίκες που γίνονται με τη νέα νομοθεσία κρατάνε λιγότερο από ό,τι προηγουμένω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικαστήρια και τη δυνατότητα να κάνουν αποτελεσματικότερη εργασία. Συνεργαζόμαστε στενά με, με τους προέδρους των μεγάλων δικαστηρίων του ε, Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα δράσης για τα δικαστήρια εκείνα που έχουν ε, πολλές παλιές υποθέσεις και δεν αποφασίζουν γρήγορα. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι να υπάρξει μια κατάρτιση των προέδρων των δικαστηρίων. Μπορεί να είναι καλοί δικαστές, αλλά δεν είναι καλοί, δι, καλά διοικητικά στελέχη, καλή διευθυντικά, καλά διευθυντικά στελέχη. Δημιουργήσαμε λοιπόν τη, ένα, μια νέα θέση, τη θέση του διευθυντή δικαστηρίων για τα δικαστήρια που έχουν ε, πολλές εκκρεμείς υποθέσεις. Και αν δεν πετύχουμε ή αν δεν πετύχει ένα δικαστήριο, αντικαθίστε το πρόεδρο του δικαστηρίου και προσλαμβάνουμε ένα νέο διευθυντή. Τελευταίο ζήτημα. Πρόγραμμα προστασία μαρτύρων. Έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Ενισχύουμε ωστόσο το πρόγραμμα με νέα στοιχεία. Το Δεκέμβριο ε, υιοθετήσαμε ένα νέο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα προστασίας των δυνάμει μαρτύρων, ατόμων δηλαδή που δεν έχουν κληθεί ως μάρτυρες αλλά που θεωρούμε ότι μπορεί να, χρησιμο... να χρησιμεύσουν ως μάρτυρες. Προσφέρουμε δηλαδή προστασία σε άτομα που μπορεί να έρθουν ως μάρτυρες μόνο και μόνο για να τους ενθαρρύνουμε. Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης της θέσης των μαρτύρων, ένα πρόγραμμα υποστήριξης των μαρτύρων ειδικότερα. ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ελπίζουμε να καλύψει όλους στο εγγύς μέλλον. Το πρόγραμμα υποστήριξης έχει ως εξής. Ένας μάρτυρας που έρχεται σε ένα ξένο περιβάλλον του δικαστηρίου. Χρειάζεται να ταξιδέψει π.χ. Υπάρχει ένα ειδικό δωμάτιο και άνθρωποι που τον βοηθούν να αισθανθεί άνετα, να προετοιμαστεί, Ψυχολογική υποστήριξη του μάρτυρα είναι αυτή δηλαδή. Και έχει καλά αποτελέσματα. Επηρεάζει τις δίκες. Στο πρόγραμμα αυτό συνεργαζόμαστε με το UNDP, με το πρόγραμμα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΙΕ και κάποιες κυβερνήσεις έρχονται και κάποιοι ειδικοί άλλοι δουλεύουν επαγγελματικά και άλλοι σε θελοντική βάση. Φοιτητέ, ψυχολογίες και τέτοια, κάνουν πρακτική. Αυτά. Κύριε Σιμόνοβιτς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισκεψή σας, για το χρόνο που μας διαθέσατε, για τις ε, ειλικρινείς απαντήσεις σας. Και όπως ε, ήδη είπατε, ή μάλλον σας είπαμε εμείς, ε, σας προσφέρουμε την αμέριστη υποστήριξή μας. Ευχόμαστε την ένταξη της χώρας σας, είναι σημαντικό και για την ίδια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή τύχη. Now, We will have short break and we will meet again. Κάνουμε τώρα διάλειμμα και θα ξανασυνθούμε στις 4.30 ε, με τις ε, ηλεκτρονικές μας ε, κάρτες γιατί θα ψηφίσουμε.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 accept Turkey to become at last voting. Encouraged by Sir Robert, I proceed to the vote. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να βάλετε την κάρτα σας στη θηρίδα. Ε, θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά της ψηφοφορίας που ξεκινάμε με την ε, έκθεση Σαντίβανη και μετά προχωράμε στη Βραζίλια της κυρίας Κοπά και μετά ε, στην απαλλαγή Σαντίβανη μετά Μπαγκέτ Κούτσεκ και στο τέλος θα ψηφίσουμε την πιο ωραία έκθεση που είναι η Τουρκία λέει χαριτολογώντας ο πρόεδρος. Turkish, Turkish Delight χαρακτηριστικά στο τέλος. Λουκούμι δηλαδή της Τουρκίας. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφορία. Uh, draft opinion on the draft uh, on the draft opinion. No. Opinion on the accession. Draft opinion on control of budgetary implementation of the instrument for pre The rapporteur Συγητής λοιπόν είναι ο κύριος Σεντίβανη. Δύο τροπολογίες, η τροπολογία υπαριθμών 1, ε, δεν ηλεκτρονικά, υπέρ παρακαλώ. Οι δύο εγκρίνεται και αυτή. Η ηλεκτρονική ψηφορία για το σχέδιο της γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και το αποτέλεσμα είναι υπέρ. Συγχαρητήρια 57-0. Ομόφωνα. Ψηφίστηκε η ε, γνωμοδότηση ομόφωνα. Τώρα πάμε σχέδιο έκθεσης με πρόταση για σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βραζιλία. Είναι η έκθεση της κυρίας Κοπά, της κυρίας Μαρίας Ελένη, Ελένη Σκοπά. Ε, υπέρ παρακαλώ. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Θέλετε να ελέγξουμε. Μετά πάμε στην 8 υπέρ. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Εγκρίνεται. 11 εγκρίνεται. 12 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Εγκρίνεται. 3 ε, υπέρ. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ Κατά παρακαλώ. Εγκρίνεται. Μία, ένα υπέρ, δύο υπέρ, τρία, εγκρίνεται συγγνώμη. Και πρέπει να ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Μπορούμε να ψηφίσουμε unblock σε, με, για περισσότερες τοπολογίες, σώματι. Έτσι λοιπόν... 3, 4, 5 από κοινού υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Και οι 3, οι 6 υπέρ απορρίπτεται. Οι 7 υπέρ εγκρίνεται. 8 υπέρ εγκρίνεται. 9 υπέρ εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης ως τροποποιήθηκε υπέρ παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία και τώρα έκλεισε και το αποτέλεσμα είναι 56 με 3 συγχαρητήρια κυρία Κοπά. Φτάνουμε λοιπόν στην ε, επόμενη ψηφοφορία, στην υπαριθμόν 3. Δεν είναι η Τουρκία, είναι και πάλι έκθεση Σαντίβανη. Πού είναι η κυρία Σαντίβανη? Draft σχέδιο γνωμοδότησης ε, ε, για το 2007 και έχουμε δύο τροπολογίες, την πρώτη υπέρ, εγκρίνεται, οι δύο υπέρ, κατά, εγκρίνουμε για την δύο, άρχεται ηλεκτρονική ψηφορία. Έκλεισε το αποτέλεσμα είναι 2631, ε, δηλαδή απορρίφθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο της γνωμοδότησης. Ως τροποποιήθηκε, ε, παρακαλώ ψηφίστε, άρχεται η ψηφοφορία, έκλεισε και το αποτέλεσμα είναι 61. Ε, συγχαρητήρια πέρασε η ε, γνωμοδότηση. Μετά πάμε στον διάλογο με τους πολίτες Ευρώπης, έκθεση Κούτσεκ. Και περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ παρακαλώ. Κατά απορρίπτεται. Η 3 υπέρ εγκρίνεται. 2 υπέρ εγκρίνεται. 5 ε, σε δύο τμήματα ψηφίζουμε, σε τρία μάλλον. Για το πρώτο τμήμα τροπολογία υπαριθμών 5 υπέρ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 6 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει. Η 13 υπέρ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. 8 υπέρ παρακαλώ. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Εγκρίνεται. 10 υπέρ απορρίπτεται. 11 υπέρ εγκρίνεται, η 12 υπέρ εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο όσο τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, έκλεισε η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα είναι 64-0. Ε, συγχαρητήρια. 64-7 είναι το αποτέλεσμα. 0 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Κούτσεκ. Και τώρα πάμε στο λουκούμι, το τουρκικό. Turkish Delight, λέει ο πρόεδρος. Το άφησα για το τέλος. Μετά από μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, τώρα θα έχουμε μια μακροσκελέστατη ψηφοφορία. Λοιπόν, να συγκεντρωθείτε στις ε, τροπολογίες ε, για να περιορίσουμε λιγάκι το μαρτύριο, όχι για την Τουρκία, αλλά για μας. Είναι μια πολύ καλή δουλειά της κυρίας Όμεν αλλά η έκθεση είναι μακροσκελής, όπως σας είπα. Παρακαλώ να είστε συγκεντρωμένοι και εγώ θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος. 21 υπέρ, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά. Εγκρίνουμε την 22, ε, ελέγχουμε την 22. Ελέγχουμε την 22. Παρακαλώ να ψηφίσετε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα 12.35 απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Απο, ε, απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 24. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έκλεισε και το αποτέλεσμα είναι 20 προς 42 απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Προφορική τροπολογία. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ. Εγκρίνεται. 24, μάλλον 25. 26 υπέρ. Απορρίπτεται. 27 και 28 από κοινού υπέρ παρακαλώ απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ εγκρίνεται. 30 υπέρ απορρίπτεται. 31 υπέρ απορρίπτεται. 33 υπέρ απορρίπτεται. 34 υπέρ απορρίπτεται. 35 υπέρ εγκρίνεται. 36 υπέρ εγκρίνεται. 37 υπέρ απορρίπτεται. 38 υπέρ απορρίπτεται. 39 υπέρ απορρίπτεται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 39 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Εδώ πρέπει μάλλον να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 39 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική 2. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Μισό λεπτό. Εγώ θα ήθελα να είμαι υπέρ αυτής της τροπολογίας, αλλά στο τέλος της παραγράφου 14 να μπει αυτή στο τέλος της παραγράφου 14. Η 42 υπέρ κατά, ελέγχουμε τη 42, άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίστε για τη 42, έκλεισε. Ε, Πάμε στην 3 υπέρ. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Απορρίπτεται. Η 46 υπέρ απορρίφθηκε. Η 48 υπέρ. Καλύπτεται. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην 53 υπέρ παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 υπέρ εγκρίνεται. Η 60 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ εγκρίνεται. Η 62 υπέρ εγκρίνεται. 63 σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα το 63 υπέρ παρακαλώ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ εγκρίνεται. 64 υπέρ απορρίπτεται 65 υπέρ εγκρίνεται 66 υπέρ απορρίπτεται 67 υπέρ απορρίπτεται 68 υπέρ απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ εγκρίνεται 70 υπέρ απορρίπτεται 72 υπέρ μισό λεπτό συγγνώμη λέει ο πρόεδρος δικό μου το λάθος 74 υπέρ απορρίπτεται. 77 υπέρ απορρίπτεται. 78 υπέρ απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ εγκρίνεται. 80 υπέρ απορρίπτεται. 81 αποσύρθηκε. 83 υπέρ απορρίπτεται. 84 υπέρ απορρίπτεται. 86 υπέρ απορρίπτεται. 87 υπέρ εγκρίνεται. 87. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 87. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λάθος έκανε ο πρόεδρος. πρώτο κανόνα είναι ο πρώτο έχει δίκιο. Δεύτερον, αν δεν έχει δίκιο, βλέπε κανόνα 1. Συμβαστική 8 υπέρ, δεκτή. 91. Απορρίπτεται. 92. Απορρίπτεται. 93. Απορρίπτεται. 94. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Δεκτή. 96 υπέρ. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Δεκτή. 99 υπέρ. Απορρίπτεται. 100. 101 και 102 παρόμοιες, ίδιες, υπέρ, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Δεκτή. 104. Όχι. Δεν με είδατε. Υπήρχε μια προφορική τοπολογία που αποσύρθηκε, αλλά μπορεί να επανέλθει στην Ολομέλεια. Δεν υπάρχει προφορική τοπολογία. Δεν υπάρχει προφορική τροπολογία. Θα υπήρχε μια πιθανή αλλαγή με βάση τις θέσεις της Επιτροπής Γυναικών. Δεν έγινε όμως αυτό σήμερα. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει ίσως πριν την Ολομέλεια. Ό,τι θέλει η συγκήτρια. 107 υπέρ. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Δεκτή. 109 υπέρ. Απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, έλεγχος για την 110. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. κάθαρα αποδείχθηκε λέει ο κύριος Γκάλερ. 112 υπέρ. 111 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Δεκτή. 113 υπέρ. 113 υπέρ. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Απορρίπτεται. 115 καλύπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Δεκτή. Καλύπτονται. 120 υπέρ. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία Βλέπει την παράγραφο 27 υπέρ. Δεκτή. Δεν ψηφίζουμε από αυτού. 125 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 125. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι. Πλήρης απόρριψη. Βοηθήστε με κύριε Γκάλερ περισσότερο. 126 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 126. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Σαλαφραγκά, η ομάδα σας έχει τρεις βουλευτές πάνω από τα όρια. Τώρα, τώρα είναι εντάξει. Δεν είναι ότι έχουμε στο παρά ένα και στο και ένα ψηφοφορίες, αλλά ζητώ από τους συντονιστές να μην ξεπερνάτε το 100% της παρουσίας. 120, όχι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ήταν 126 κάναμε. Αρχίζει ξανά η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Με αποτέλεσμα. Απόρριψη. Απορρίπτεται 126. 127 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 127. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Δεκτή. 130 υπέρ. Δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ ναι, ναι. Ναι, κύριε Λαμστόφ. Εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, έχουμε μία προφορική τροπολογία στην συμβαστική πρόταση 11. Η φιλελεύθερη ομάδα πιστεύει ότι η ελευθερία της συνέλευσης ε, και το ε, δικαίωμα διαδήλωσης θα πρέπει να ισχύουν 365 μέρες το χρόνο και σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο την 1η Μαΐου και στο Ταξίμ. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνουμε αυτό που κάνει λόγο το Ταξίμ να αφαιρεθεί και να προβάλλεται στο σύνολό είσαι η ελευθερία αυτή. Παρακαλώ λοιπόν οι συνάδελφοι να στηρίξουν αυτή μου την τροπολογία. Κοιτάξτε, το καλύτερο από όλα θα ήταν τότε να έχουμε ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτα θα ψηφίσουμε για το σύνολο του κειμένου χωρίς αυτή την πρόταση και μετά ο καθένας θα αισθάνεται ελεύθερος να ψηφίσει όπως θέλει. Λοιπόν, να κάνουμε το εξή, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε πρώτα για το κείμενο με διαγραφή, διαγράφοντας όλο αυτό το κομμάτι που λέει την 1η Μαΐου στο Ταξίμ, στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς αυτό το κομμάτι. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ του κειμένου με διαγραφή αυτού που σας είπα, εντάξει. Ε, δεν έχει κανένα νόημα να επαναλάβουμε. Έτσι λοιπόν η συμβαστική 11 εγκρίνεται χωρίς... Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό πρέπει να ψηφίσουμε τώρα και για το να ενταχθεί αυτή η πρόταση. Έχετε δίκιο κύριε Λάμστορ. Λοιπόν, θα αποφασίσουμε τώρα κατά πόσο θα προσθέσουμε αυτή την πρόταση που λέει 1η Μαΐου Ταξίμ. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Ως εκ τούτου, οι διαδηλώσεις θα γίνονται στην Τουρκία την 1η Μαΐου, στην πλατεία Ταξίμ. 134 υπέρ απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κύριε Λάμπστοφ, τι θέλετε. Κοιτάξτε, στην ε, ε, συμβαστική πρόσθεση θα πω στα αγγλικά. Έχουμε μια προφορική τροπολογία για την 12 που αναφέρεται στη ε, γραμμή στο τέλος που λέει καλεί την Τουρκία να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα. Αυτό θέλουμε να το τροποποιήσουμε και θα λέει καλεί την Τουρκία να διευκολύνει ευνοϊκό κλίμα για διαπραγματεύσεις ξεκινώντας την απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων. Πιστεύουμε ότι το να γίνει η πλήρης απόρριση των στρατευμάτων για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτό είναι παντελώς ουτοπικό. Εκεί σημαίνει ίσως ότι τελειώνει όλη η διαδικασία. Όπως ήδη είπα το πρωί στη συνεδρίαση, είπα ότι η απόσυση τουρκικών δυνάμεων δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποσυρθούν όλες. Καλύπτει η συμβιβαστική μου πρόταση όλα όσα επιθυμείτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να αλλάξουμε το συμβαστικό κείμενο. Κύριε Σβόμποντα, να παραμείνουμε στην ερμηνεία της εισηγήτριας, οπότε ψηφίζουμε την ε, τροπολογία της συμβαστική ως έχει. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε λοιπόν τη διατύπωση, την πρωτότυπη, την αρχική, συμβιβαστική 12. εισηγείται είναι κατά, οπότε δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την προφορική τροπολογία. Αυτό είναι ο κανόνα. Η κυρία Μεν Ράιτν. Για να του κάνω χάρη, μπορούμε να ψηφίσουμε όλο το κείμενο και αν θέλει αλλαγή από αυτού μπορούμε να ψηφίσουμε μετά. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Είμαστε πολύ συμφιλιωτικοί. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο ως παρουσιάστη υπέρ. Εγκρίνεται και τώρα ποιος είναι υπέρ της αντικαταστάσεως της αποσύσεως με την έναρξη της αποσύσεως. Παραμένει το αρχικό κείμενο, αρχική διατύπωση. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 12 υπέρ. Εγκρίνεται 135 υπέρ. Πρέπει να πάτε στην αρχική ψηφοφορία κατά τμήματα, λέει ο Σλάγκεντάικ. Για τις τέσσερις ελευθερίες. Δεν ψηφίσαμε τις τέσσερις ελευθερίες ψηφίσαμε την πρόταση του Άλεξ. No, there is a split vote. Take... Κατά τμήματα σου φορεί αναφέρεσαι τις λέξεις συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών. Είμαι υπέρ όλου του συμβιβασμού, αλλά θέλω αυτέ οι λέξει να διαγραφούν και θέλω να το ψηφίσουμε αυτό που προτείνω εγώ. Ψηφίσαμε, λέει η κυρία Όμεν Όχι, έρχεται η απάντηση. Ψηφίσαμε, λέει η κυρία Όμεν Ψηφίσαμε, αλλά it's not fair to me. You, you put to the vote the whole chemical issue. In his first part. Yes, but the first part Okay, to make, to make the things clear. Για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία συμβαστική 12, πρώτο τμήμα Όλος ο συμβιβασμός εκτός από τις λέξεις συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών. που είναι υπέρ. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Δεύτερο τμήμα. Με αυτές τις λέξεις υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στα 135 υπέρ. Απορρίπτεται. is compatible. Είναι συμβατή η 135 δεν καλύπτεται αλλά είναι συμβατή 135 απερίφθη. Πάμε στην 139 υπέρ. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 145 υπέρ. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. I'd like to... Uh, Πρόεδρε, θέλω να αποσύρω την 149, λέει και ο Μιλανδένοφ. Αποσύρεται την 149 ήταν της κυρίας Νίκολσον. Λοιπόν, 149 απορρίπτεται. Η Βαρόνι Νίκολσον δεν αποσύρει. Ο κύριος Μλαντένοφ μπορεί να αποσύρει τη δική του τροπολογία, αλλά όχι η Βαρόνι Νίκολσον. Μόνο το μισό ψηφίζουμε, λέει, τη μισή τροπολογία Ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Ποιο, το πρώτο ή το δεύτερο μισό. αν και οι δύο δεν αποσύρουν, ψηφίζουμε την 149 υπέρ, κατά, απερίφθη, 150 υπέρ, εγκρίνεται, 151 υπέρ, απορρίπτωται 153 υπέρ, απορρίπτωται 154 υπέρ, κατά, έλεγχος της 154. Ξεκινάνε τη ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας 154. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Συμφωνείτε. Σημειώνουμε αυτό που μας λέτε. 155 υπέρ. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 157. Ξεκινάμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι απόρριψη 31 με 33 απορρίπτεται με μικρή διαφορά Πάμε στην 158 υπέρ. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Απορρίπτεται. 160 καλύπτεται. 161 αποσύρεται. 162 υπέρ. Κατά έλεγχος της 162. Ξεκινάμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Και το αποτέλεσμα είναι απόρριψη. 163 υπέρ απορρίπτεται 164 υπέρ απορρίπτεται 165 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα της 165 υπέρ κατά απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ εγκρίνεται 166 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ απορρίπτεται 167 168 υπέρ κατά έλεγχος για την 168 ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίστε παρακαλώ τέλος ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα έχει ως εξής 35-34 άρα εγκρίνεται με διαφορά μιας ψήφου είναι σωστή αριθμή των μελών δεν περισσεύει κάποιος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 Τρίθηκε η ψήφο σας. 169 υπέρ. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. θα ελέγξουμε την 170. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα. 23 με 44 και απορρίπτεται η 170 δεν σηκώνεται τα χέρια καλά 171 υπέρ κατά έλεγχος για την 171 ξεκινάμε ψηφίστε παρακαλώ πέρα ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι απόρριψη ευχαριστώ κύριε Γκάλερ 172 172 υπέρ απορρίπτεται 173 υπέρ απορρίπτεται 174 υπέρ. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Εγκρίνεται. 178 υπέρ. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Απορρίπτεται. 181 υπέρ. Εγκρίνεται. 182 υπέρ απορρίπτεται. 183 υπέρ, απορρίπτεται. 184 υπέρ, απορρίπτεται. 185 υπέρ, απορρίπτεται. 187 υπέρ, απορρίπτεται. 188 υπέρ, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, εγκρίνεται. Καλύπτονται, καλύπτονται, καλύπτονται. 12 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Δεν αποσύρεται 15. Λοιπόν υπέρ της 15. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Έλεγχος της 18, ηλεκτρονική ψηφοφορία 18, ηλεκτρονικός έλεγχος, πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι απόρριψη. Με διαφορά 7 ψήφων. Προφορική τροπολογία της αιτιολογικής εφλατινικό υπέρ εγκρίνεται. 19 υπέρ απορρίπτονται. 20 υπέρ κατά Έλεγχος της 20, ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει, πέρα ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι απόρριψης. Ένα υπέρ, η Ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική για το λουκούμι μας, για την Τουρκία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ και το αποτέλεσμα είναι θετικό. 65 με 4 με μία αποχή. Συγχαρητήρια Μεν Ρόιτεν. Πολύ καλή δουλειά. Η ε, κυρία Μεν Ρόιτεν έχει κάτι να μας πει. Είχε το λόγο. Ναι, λέει η κυρία Μεν Ρόιτεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν για αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, ε, επίσης και όλους τους βοηθούς μάλλον όλη τη βοήθεια που πήρα, όχι μόνο από την ΕΒΑ, από τη γραμματεία της Επιτροπής, από τη γραμματεία του ΕΛΚ, από τους βοηθούς μου. Χάρη σε αυτούς πέρασαν οι δύσκολες εβδομάδες και έφτασα αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζω να δώσει νέα όθηση στην Τουρκία. Είναι δίκαιη η έκθεση, ειλικρινής, αλλά θα πρέπει να δείξουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ τους πάντες, ευχαριστεί η Επιτροπή, την κυρία Ομεν και την ομάδα της. Πέρα στη συνεδριά σα σας ευχαριστώ.